Αγαπητοί συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε. Τρεις και πέντε η ώρα πια. Καλώς ορίζω τους 30 επισκέπτες μας. Μια ομάδα προσκεκλημένη του φιλελεύθερου κόμματος, του κόμματος των φιλελευθέρων στη Γερμανία και του Πέτερ Ράιμερ συγκεκριμένα. Καλώ ήρθατε στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να σα φανούν ενδιαφέρουσε οι συνομιλίες. Θα παρατηρήσετε πρώτα-πρώτα ότι πλην του κυρίου Καντσάν οι βουλευτές από τη Βόρεια Ευρώπη έρχονται εγκαίρω, προσέρχονται εγκαίρως συνεδρίε, ενώ εκείνοι της Νότιας Ευρώπης τείνουν να τραβάνε το χρόνο λίγο περισσότερο. Και γι' αυτό ξεκινάμε με πέντε λεπτά καθυστέρηση. Καλώς ήρθατε πάντως. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η έγκριση του σχεδίου. Είμαστε όλοι σύμφωνοι, πολύ καλά. Δεύτερο, η έγκριση των πρακτικών της 30ης Ιανουαρίου, της 10 Φεβρουαρίου και της 20ης Φεβρουαρίου. Δεν υπάρχουν προβλήματα και περνώ στο επόμενο και τρίτο θέμα. Πρόσβαση στην αγορά λιμενικών υπηρεσιών και χρηματοοικονομική διαφάνεια των λιμένων, κανονισμός, ανταλλαγή απόψεων. Ξέρετε ότι η αυριανή ψηφοφορία έχει αναβληθεί. Ο κύριος Φλέκινστάιν με την παρουσίαση του θέματος θα μας εξηγήσει γιατί έλαβε την απόφαση αυτή ο πρόεδρος. Κνούτ, έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε εδώ να κάνουμε με ένα κανονισμό που εσφαλμένο ονομάζεται τρίτο πακέτο για τα λιμάνια που δεν είναι καθόλου εύκολη δουλειά για μας. Είχαμε μια μήνυα ακρόαση με βρετανικά, φινλανδικά ε, λιμάνια, τη, Μασαλία, το Ρότερνταμ ε, και ανταλλαγή απόψεων με λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς στην ΕΣΠΟ, με τους εφοπλιστές, ε, συνδικάτα κτλ. Έχουμε στο πλαίσιο αυτών των διαβουλεύσεων ε, καταλήξει σε κάποιες συμβαστικές λύσεις ε, στην συνεργασία μας με την Επιτροπή, στη διαφάνεια, στο περιθώριο χειρισμών, τις δυνατότητες περιορισμού των, του αριθμού των ε, φορέων παροχής υπηρεσιών, το, τις κοινωνικές, ελάχιστες κοινωνικές προδιαγραφές, το κατάλογό μας και ιδέες όπως ε, αποφυγή της γραφειοκρατίας στο, στο δυνατό για τους ελέγχους και την λήψη των αποφάσεων και έτσι θα ήθελα να ευχαριστώ θερμά τους εκπροσώπους των Γενικών Διευθύνσεων ε, της Επιτροπής για την πολύ καλή συνεργασία. Πάντως, τελευταία εβδομάδα, στην εβδομάδα στο Στρασβούργο, διαπιστώσαμε ότι δεν είμαστε σε θέση να κλείσουμε τον κανονισμό αυτόν και να τον εγκρίνουμε στο πλαίσιο της θητείας μας. Για δύο λόγους. Καταρχάς, διότι δεν έχουμε καταλήξει σε συμβασμό προς το πεδίο εφαρμογή του κεφαλαίου για την πρόσβαση στην αγορά, γιατί η Επιτροπή έχει διαγράψει τα κομμάτια που αφορούν τα δικαιώματα των ε, ε, επιβατών και επίσης διότι δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν οι ομάδες. Έτσι λοιπόν η απουσία στα δύο αυτά θέματα που αποτελούν και την ουσία του κανονισμού δεν μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στα τυφλά και να αφήσουμε στην τύχη την έγκριση του θέματος. Επίσης έχουμε επισημάνει ότι θα πρέπει τον, τον κανονισμό αυτό να τον βλέπουμε πάντοτε σε συνεργασία με τις ε, σχετικές με τις διατάξεις σχετικές με τις ε, αναθέσεις και την παροχή των υπηρεσιών ε, στους λιμέν, στις, με κρατικές επιδοτήσεις. Δεν μπορέσαμε όμως να συμφωνήσουμε σε μια κοινή εικόνα και έτσι κάναμε σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση για τον Ανταγωνισμό αλλά και για τις μεταφορές μία στην συζήτηση. Στους δύο τομείς παραμένουν οι ανησυχίες μας, αφενός μεν οι ε, διατάξεις για τις ενισχύσεις της υποδομές, όπου ισχύουν ε, κατευθύνες γραμμές που δεν έχουν ε, υποβληθεί πιο πριν και οι, εξα... οι εξαιρέσεις όπου για τις υποδομές δεν προβλέπουν ειδικού κανόνες. μπορεί από το 2015 να αρχίσει να ισχύει, αλλά αμφιβάλλουμε εάν θα υπάρξουν αποφάσεις, γιατί έχουμε πολύ λίγες μέχρι τώρα αποφάσεις δικαστηρίων που να ρυθμίσουν τα θέματα αυτά. Επίση το ερωτηματολόγιο, τα ερωτηματολόγια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή που απευθύνονται σε διάφορα κράτη μέλη σε σχέση με τον εταιρικό φόρο, είναι ένα άλλο ζήτημα συνάντησή μας με την Επιτροπή και τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού είχε σαν στόχο να κοιτάξουμε γιατί έχει αναβληθεί αυτό το θέμα. Δεν λάβαμε όμως καμία λογική απάντηση. Και επίσης μας απασχολεί το θέμα της γενικής ρύθμισης των επιχειρήσεων στα λιμάνια, το, τα πουλ αυτά όπως ονομάζονται, με τον κίνδυνο να μπουν από την πίσω πόρτα, όπως φοβόμαστε, κάποιες ρυθμίσεις από την Επιτροπή. Και έτσι είπαμε ότι είναι καλύτερο να επεξεργαστούμε περαιτέρω τα θέματα, ώστε να ξέρουμε επακριβώ τι έχει υπόψη η Επιτροπή Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού. Απέστειλα λοιπόν επιστολή στον πρόεδρο της Επιτροπής μας, τον Brian Simpson, του εξήγησα ποια είναι η κατάσταση, πόσο έχουν προχωρήσει οι συμβασμοί και όπως το είπε και μια επιστολή στην Επιτροπή από πλευράς του και έτσι η νέα Επιτροπή Μεταφορών θα χρειαστεί οπωσδήποτε να ασχοληθεί με το θέμα αυτό διότι δεν μπορεί νομίζω η Επιτροπή να πει ότι δεν χρειάζονται όλα αυτά και ότι επί 10 χρόνια που ασχολούμαστε με το θέμα κάναμε λάθος. Άρα λοιπόν προχωρούμε με την επόμενη θητεία με πιο ασφαλή βήματα ελπίζω και πιο γρήγορα. Και φαντάζομαι ότι και η Επιτροπή θα λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις που εντυπωθούν και σήμερα. Και ελπίζω να μην χρειαστεί να ε, ανοίξουμε πανιά για να κλείσουμε τα θέματα πολύ βιαστικά ε, στο τέλος της θητείας. Ο κύριος Δεμπάκερ, φιλελεύθερη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο κύριος ε, Φλέκενστάιν σε γενικές γραμμές. Εδώ και αρκετές εβδομάδες μιλούσαμε για την ε, πρόταση της Επιτροπής. Η αρχή ήταν πολύ καλή, αλλά στη συνέχεια την, ε, τις τελευταίες εβδομάδες προσπαθήσαμε να οργανώσουμε ακροάσεις, να έρθουμε σε επαφή με την Επιτροπή, όχι μόνο την σχετική Γενική Διεύθυνση, αλλά και άλλες υπηρεσίες της Επιτροπής έτσι ώστε να υπάρχει διαφάνεια. Αλλά στο τέλος δεν προέκυψε διαφάνεια σε αυτή τη σύντομη χρονική περίοδο. Εν ώψη των εκλογών δεν μπορούμε να ικανοποιηθούμε και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να ορίσουμε καλύτερα την πρόταση, να την οριοθετήσουμε καλύτερα ως προς τις ε, ε, εμπορικές δραστηριότητες τους λιμένες για να προχωρήσουμε. Αλλά το άνοιγμα της αγοράς και η προσβασιμότητα της αγοράς σε αυτά τα δύο θέματα δεν βρήκαμε συμβασμό. Είναι πολύ κρίμα, αλλά έτσι έχει η κατάσταση. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε μία πρόταση και μία ε, σαφή οριοθέτηση για, τις, ε, για την πολιτική μας τους λιμένες. Πρόκειται για στοιχεία ζωτικής σημασίας έτσι ώστε να υπάρξει και νομική διαφάνεια για την εσωτερική ε, ανταγωνιστικότητα ή τις σχέσεις ε, μεταξύ λιμένων. Θα πρέπει να δούμε ποιες επιδοτήσεις γίνονται που διασαλεύουν την τάξη καθώς και τον κοινωνικό διάλογο. Θα πρέπει να υπάρχει σαφήνεια για το μέλλον και διαφάνεια. Από πλευράς της δικής μου ομάδας λοιπόν μπορούμε να αναπέμψουμε αυτό το θέμα το οποίο θα είναι ένα θέμα προτεραιότητα στην επόμενη θητεία για την Επιτροπή Μεταφορών και ελπίζουμε να φτάσουμε σε μια καλή, σε έναν καλό συμβασμό, σε μια καλή συμβιβαστική λύση για τους κανόνες οι οποίοι είναι απαραίτητοι για να υπάρχει νομική ασφάλεια για όλους τις ε, λιμένες. Αυτό ήδη υπογραμμίστηκε. Οι λιμένες αποτελούν τη σπονδυλική στήλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να, υπάρχουν, ε, να υπάρχει αρκετή ευελιξία έτσι ώστε να κρατήσουμε αυτή την ευημερία και για το μέλλον. Κύριο Κράμερ, είναι η τρίτη φορά που έχω να ασχοληθώ με το πακέτο για τους λιμένες. Πριν από 10 χρόνια που εξελέγησε το Κοινοβούλιο, το Κοινοβούλιο στην προηγούμενη του σύνθεση με την κυρία Λοιόλαντε Παλάσιο, που ήταν τότε επίτροπος αρμόδια για τις μεταφορές, είχε να εξετάσει αυτή την πρόταση που υποβλήθηκε την Επιτροπή, την ανέπεμψε το Κοινοβούλιο και χωρίς να αλλάξει το παραμικρό στο κείμενο αυτό, επανέρχεται το θέμα αυτό ε, περίπου έξι μήνες αργότερα. Ο κύριος Γιαζεμπόφσκι από το, από το Αμβούργο και πολλοί άλλοι ε, ε, αντέδρασαν, αντιδράσαμε έντονα Απερίφθη το πακέτο και πάλι και τώρα βλέπουμε να ξαναγυρίζει. Αλλά φαίνεται ότι δεν σταματάει τι προσπαθίε τη Επιτροπή. Και έτσι η κατάσταση είναι εξή, ότι κάνει αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων για λιμένε η Επιτροπή. Και έρχεται ταυτόχρονα να προτείνει νέα νομοθετήματα. Πράγμα το οποίο είναι παράλογο. Είτε γίνεται αναθεώρηση των κρατικών ενισχύσεων και εξηγούμε τι κάνουμε, είτε ξεκινάμε την πρωτοβουλία για τα λιμάνια και έτσι κλείνει η υπόθεση. Θυμάμαι και το ε, και την αναθεώρηση 1370, 1370 με τις ε, προτάσεις πάλι για τους ε, σιδηροδρόμους, με προτάσεις που ήδη είχαν τεθεί σε ισχύ στη Γερμανία και ερχόταν η Επιτροπή να αναθεωρήσει. Ε, πράγμα το οποίο δείχνει ότι η Επιτροπή ούτε καν κοιτάει τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι εφαρμόζεται, πού υπάρχουν προβλήματα, πού χρειάζεται τροποποίηση. Απλώ έρχεται και καταθέτει προτάσει. Μια Επιτροπή λοιπόν που έχει τόση εμπειρία και που στην ίστατη στιγμή έρχεται σε ένα θέμα τόσο, με τόσο βεβαρημένο ιστορικό όπω αυτό των λιμένων να καταθέσει τι ίδιε προτάσει. Ε, εμένα με ξεπερνά και πολιτικά ακόμα δεν αντιλαμβάνομαι πώς το κάνετε αυτό. Έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία στο θέμα αυτό. Γιατί λοιπόν καθώς ήσταν τέσσερα χρόνια σε κατάσταση ύπνωση, σκέφτεσαι και σε τελευταία στιγμή να μας καταθέσετε τέτοιου είδους προτάσεις. Μην ε, ξαφνιάζεστε λοιπόν αν απορριφθεί αυτό. Και θα κάνετε και το ίδιο πάλι φαντάζομαι. Στην προσεχή θητεία θα περάσουν πέντε χρόνια και πάλι θα περιμένετε μέχρι ότου την τελευταία στιγμή καταθέσετε ναι, τις ίδιες προτάσεις. Τι θέλετε λοιπόν να αποφασίσετε. Θέλετε αναθεώρηση των ενισχύσεων, κρατικών ενισχύσεων για τους λιμένες ή νέο νομοθέτημα ή μήπω τελικά θέλετε να κοιτάξετε και να αναλύσετε την πραγματικότητα, πράγμα το οποίο πράγματι είναι απαραίτητο και γρήγορα. Κύριος Bradburn, Ευχαριστώ. Πρέπει να πω ότι για πρώτη φορά θα συμφωνήσω πλήρως με τον κύριο Κράμερ. Μήπως έχω κάνει κάποιο λάθος, λέει ο κύριος Κράμερ. Ναι, Επιτέλους, μία φορά τα τελευταία πέντε χρόνια συμβαίνει αυτό και ε, πραγματικά συμφωνώ με τις απόψεις του για την ε, αποτελεσματικότητα του να φέρουμε αυτές τις προτάσεις σε αυτή τη φάση, αφού δύο φορές απορρίψαμε προτάσεις από την Επιτροπή προηγουμένως. Και βέβαια δεν είναι μόνος ο κύριος Κάμερ, εσείς και εγώ, Πρόεδρε, ήμασταν εδώ όταν ε, περάσαμε τις πρώτες δύο απόπειρες και ωστόσο όπως είπα και στην αρχή αυτή της συζήτησης, στην αρχή του χρόνου δεν μπορούμε να λέμε δύο φορές όχι και η Κομισιόν να επανέρχεται με μια άλλη δέσμη ε, νομίζοντας ότι θα αλλάξουμε γνώμη. Είναι σαφές ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις που είχαμε τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες δείχνουν ότι ο κανονισμός για τις λιμενικές υπηρεσίες δεν είναι εφικτός. Η Κομισιόν θα έπρεπε να το είχε σημειώσει μέσα στη συζήτηση και να είχε αποσύρει εντελώς την πρότασή της, διότι παρά κάποιες βελτιώσεις που έχουν γίνει στο κείμενο, ο κανονισμός είναι πολύ περιοριστικός. Περιορίζει ε, την ελευθερία διαφόρων διαφορετικών θαλασσιών λιμένων και λιμένων. Κάθε λιμένα είναι μοναδικό και πρέπει να λειτουργεί με ξεχωριστό τρόπο. Δεδομένου βέβαια ότι συμμορφώνεται με τον νόμο περί ανταγωνισμού και δεν πρέπει να φοβόμαστε ε, ε, ε, σε αυτή την στρατηγική που πρέπει να ακολουθούν τα λιμάνια. Αυτός ο κανονισμός διακυβεύει την ανάπτυξη τώρα που τη χρειαζόμαστε, τώρα στα συγκεκριμένα στοιχεία και λεπτομέρειες. Νομίζω έχουμε συμφωνήσει να μην προχωρήσουμε με την ψηφοφορία σε αυτή την θητεία. Για διάφορους λόγους, ε, τους οποίους ανέφερε και ο ίδιος ο ε, εισηγητής για τις κρατικές ενισχύσει. Είχαμε μια συνάντηση με τον αρμόδιο της Κομισιόν. Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια προτού προχωρήσουμε σε αυτό. Ε, συνέντηση των σκιωδών ε, περισσότερο τα πράγματα κατά την άποψή μου και δεν διευκρίνησε τα πράγματα. Και η Κομισιόν θα πρέπει να προσέξει την γενική ανησυχία σε αυτό το θέμα δεν είναι μόνο το θέμα των κρατικών ενισχύσεων. Ε, είμαστε πολύ μακριά από την συμφωνία στο πεδίο εφαρμογή του κανονισμού. Μιλάμε για την πλοήγηση, τη ρημούλκηση και πολλά άλλα σχετικά θέματα, όπου υπάρχουν εντελώς δισταμένες απόψεις σε αυτό το σώμα και όπου η δυνατότητα να έχουμε ανταγωνιστικές τιμές και να ακολουθούνται ε, μεμονωμένες στρατηγικές είναι το κλειδί στη λειτουργία των λιμένων και δεν αναγνωρίζονται ε, μέσα στη διατύπωση αυτού του κανονισμού. Κλείνοντας, Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι καλωσορίζει το γεγονός ότι δεν θα προχωρήσουμε με την ψηφοφορία σε αυτή τη θητεία του Κοινοβουλίου και επαναλαμβάνω ότι θα ήθελα η Κομισιόν να αποσύρει αυτή την πρόταση και αν δεν μπορεί να επανέλθει με μια λογικότερη, τότε θα πρέπει να αφήσουμε αυτό το θέμα να, μην το προχωρήσουμε καθόλου. Ο κύριος Ρίκε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να πω ότι ε, δεν εκφράζομαι εξ ονόματος του ΕΛΚ, το οποίο επιφυλιάσετε, αλλά προσωπικά. Θα ήθελα να κάνω δύο σχόλια γενικής υφής. Βλέπουμε την πολύ μεγάλη δυσκολία που υπάρχει να φτάσουμε σε ένα γενικό ρυθμιστικό πλαίσιο, όπως ήδη εκφράστηκε έμεσα από τον κύριο Μπραντμπερν δηλαδή τα ε, ειδικά στοιχεία, τις γεωγραφικές δηλαδή οι ιδιαιτερότητες με τις οποίες πρέπει να συμβαδίσουμε. Καταλαβαίνετε ότι τα λιμάνια διαφέρουν, ε, δεν ε, προσφέρουν τα ίδια καταφύγια, τις ίδιες δυνατότητες ελιμενισμού δεν έχουν τις ίδιες ε, ρυθμίσεις, συνεπώς δεν μπορεί το ρυθμιστικό πλαίσιο να ε, τους θέσει, να τους θεωρήσει ίσους. Είναι πολύ πιο εύκολο να βρίσκεται κανείς στη Βόρειο Θάλασσα παρά στη Μαύρη Θάλασσα από γεωγραφικής πλευράς. Άρα δεν μπορούμε να γενικεύουμε. Τη στιγμή όπου πραγματικά προσπαθούμε μέσω αυτού του νέου κανονισμού να ρυθμίσουμε την κατάσταση, αυτό σημαίνει ότι ανοίγουμε την πόρτα στον ανταγωνισμό και την ίση πρόσβαση στους λιμένες για μια πολιτική ανταγωνισμού. Και μπορούμε να πούμε ότι οι πλειοκτήτες ε, είναι το, αντίπολο, το αντίπαλο δέος ε, των, ε, στους λιμένες. Και δεν ξεχνάμε ότι ως προς τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων που αποτελούν ένα ε, μείζον μέρος της δραστηριότητας, μια δραστηριότητα που ένα και δύο διονγκούται, υπάρχει μια, ε, ένας παγκόσμιος συγκεντρωτισμός, διότι οι πλειοκτήτες ομαδοποιούνται σε τρία-τέσσερα ε, σε τρία-τέσσερα καρτέλ δηλαδή οι πρώτοι παγκοσμίω πλειοκτήτες που μεταφέρουν εμπορευματοκιβώτια ε, un très important changement dans l'offre de transport μας ε, δίνουν τη δυνατότητα να τους ομαδοποιήσουμε και δεν νομίζω ότι αυτή η κίνηση από πλευράς ε, πελατών είναι μια οργάνωση που μπορούμε να προτείνουμε μέσα στα πλαίσια μιας γενικότερης ρύθμισης. Συμφωνώ δηλαδή με τους προλαλήσαντες ότι ίσως ε, στην επόμενη θητεία θα πρέπει να γίνει μια διαφοροποίηση και ορισμένες τροποποιήσεις του νέου ε, κειμένου νομοθετικού περιεχομένου. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάισνερ. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα που ανάβει τα αίματα αυτό το πακέτο για τα λιμάνια. Στην προηγούμενη θητεία δεν προχώρησε. Στην ε, τωρινή περιμέναμε, περιμέναμε, περιμέναμε να έρθει ένα πακέτο, να έρθει ένας κανονισμός για να βελτιωθεί η κατάσταση στους λιμένες. Και από τη Γερμανία που μπορώ να, να γνωρίζω καλύτερα, ε, εκπρόσωποι είχαν πει ότι χρειάζεται μια ρύθμιση. Ε, ήρθε εν τέλει, έστω όντως πάρα πολύ αργά, αλλά από την άλλη πιστεύω ότι μπορεί να υπάρχει δυνατότητα να συμφωνήσουμε. Δεν βλέπω τα πράγματα τόσο ριζικά όπως ο κύριος Ρέντμπερν ή ο κύριος Κράμερ που λένε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι, που λένε ότι δεν ε, μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Όχι, νομίζω ότι πρέπει να κοιτάξουμε πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις προτάσεις αυτές. Βεβαίως μπορεί να υπάρχουν διαφορετικές απόψεις, αλλά έχουμε και τη δυνατότητα να κοιτάξουμε τι μπορεί να ισχύει γενικά ε, για την ε, διακίνηση φορτίων μέσα από τα λιμάνια της Ευρώπης, τι μπορεί να ισχύει γιατί επί παραδείγματι προβλέπουμε ένα σχέδιο ασφάλειας για τους λιμένες, γιατί διευκολύνουμε τις επενδύσεις, διαφυλάσσοντας όμως και τη δυνατότητα για τον ανταγωνισμό. Ε, αυτές οι πτυχές δηλαδή και των ε, της ε, διακίνησης με ασφαλή τρόπο των ε, φορτίων αλλά και των δημοσίων προμηθεών είναι κάτι που μπορούμε να συζητήσουμε. Είχε δίκαιο η Επιτροπή στο ότι έχουμε πολύ μεγάλο αριθμό φορτίων, πολύ μεγάλο όγκο διακίνηση από τα λιμάνια μας και ο κύριος Φλέκεστάιν νομίζω βλέπει ότι υπάρχει ανάγκη και αρρύθμιση. Έχει δει πολύ σωστά, ότι, γιατί κάναμε μαζί και τις ακροάσεις, ότι πρέπει να υπάρχει υποστήριξη ε, της ε, δραστηριότητας των λιμένων μας στην Ευρώπη σε αυτό συμφωνώ, έστω και αν διαφωνούμε στα υπόλοιπα, για τις κρατικές ενισχύσεις. Είμαστε στην Επιτροπή Μεταφορών. Είχαμε προσπαθήσει να εντάξουμε το θέμα αυτό και στις αρμοδιότητες του Επιτρόπου ε, του Αρμοδίου για τις Μεταφορές. Δυστυχώς δεν τα καταφέραμε. Πάει σε, άλλο, σε άλλη υπηρεσία και σε άλλο επίτροπο το θέμα αυτό, αλλά παρόλα αυτά Είμαι βεβαίω ότι θα καταλήξουμε σε μια συμφωνία, δεν αισθάνομαι ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Από την άλλη, ο κύριος Φλέκενστάιν πολύ σωστά λέει ότι δεν μπορούμε στο γόνατο να το λύσουμε. Ε, χρειάζεται περισσότερο χρόνο, ούτε καν τριμερή διάλογο δεν μπορούμε να πούμε ότι θα περιμένουμε κάποια πρόοδο. Στην επόμενη θητεία λοιπόν θα γίνει η επανεξέταση του θέματο και είμαι βεβαία ότι μπορούμε να προχωρήσουμε. Δεν, χρειάζεται να μείνει το πράγμα όπω έχουν. Πρέπει να δώσουμε μια νέα ζωή στους λιμένες μας. Κύριος Αλχαντράουι. Eh, Εκ μέρους ε, της δικής μου ομάδας θα ήθελα να συμφωνήσω με την πρόταση του κύριου Φλέκενστάιν έχει κάνει εξαιρετική δουλειά και πιστεύω ότι η Κομισιόν έσφαλε γιατί ξεκίνησε αυτό το πολύ ευαίσθητο φάκελο τόσο αργά. Δύο φορές ήδη προσπαθήσαμε να συντάξουμε μια οδηγία σε αυτό το θέμα. Θυμάμαι το 2009 η Κομισιόν πρότεινε ότι θα, θα υπήρχαν κάποιες κατευθυντήριες γραμμές σε ό,τι φορά τον κοινωνικό διάλογο και για το πώς θα οργανωνόμασταν σε αυτό τον τομέα, αλλά τελικά περιμέναμε. Ε, δεν είχαμε τα αποτελέσματα ε, και ο διάλογος να ξεκίνησε κάπως, αλλά δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει. Τον περασμένο μήνα Ακούσαμε ότι οι ενδιαφερομένοι φορείς δεν ε, ε, ήταν πολύ ευχαριστημένοι με την μικρή πρόοδο που επιτελέστηκε. Και το συμπέρασμα ήταν ότι είναι πολύ δύσκολο να τύχει διαπραγμάτευση μια τέτοια οδηγία για τις ε, λιμενικές υπηρεσίες ε, αν δεν μπορούμε να έχουμε μια καλύτερη επισκόπηση άλλων θεματών πολιτικής που έχουν να κάνουν με τα λιμάνια, για παράδειγμα τις παραχωρήσει. Θα πρέπει να έχουμε καλύτερη οργάνωση των λιμένων, αλλά μέχρι να έχουμε μια καλύτερη εικόνα της όλης κατάστασης θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια βιώσιμη λύση. Ελπίζω να καταλήξουμε σε κάποια αποτελέσματα τους επόμενους μήνες. Ελπίζω να έχουμε κάτι επιτάπητος, ε, κάποιου είδους οδηγία που θα μας ε, δώσει κάποιο υλικό ε, το οποίο να επεξεργαστούμε έτσι ώστε να βοηθήσουμε τα λιμάνια να αναπτυχθούν. Αλλά το συμπέρασμα είναι ότι από αυτές τις περιστάσεις και δεδομένων των εκκρεμουσών ερωτήσεων και θεμάτων και του περιορισμού του χρόνου, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσουμε. Θα πρέπει να περιμένουμε. Thank you very much for my... Ευχαριστώ πολύ από δικής μου πλευράς, επειδή ήμουνα σε επαφή με τον εισηγητή. Ξέρω ότι και ο κύριος Κομουτσάκος έχει την ίδια άποψη με τις απόψεις που εκφράστηκαν εδώ από τους βουλευτές. Σε αυτή τη συζήτηση γι' αυτό ε, δεν θα γίνει ψηφοφορία. Όπως ε, εισηγήθηκε και ο συντάκτης και η σκιώδης. Ο Μάικλ το ανέφερε αυτό και ο Φίλιπ το υποστήριξε όταν δει κανείς ε, την νομοθετική πρόταση ή τις νομοθετικές προτάσεις που ανέκυψαν τους τελευταίους έξι μήνες, πρόκειται για ένα μεγάλο, μακρύ κατάλογο. Ε, σιδηροδρομική, σιδηροδρομικά, ε, θαλάσσιες μεταφορές, ενίος ευρωπαϊκός ουρανός, βαριά οχήματα, ε, δοκιμές, ε, κανονισμός 261 για τα δικαιώματα των επιβατών και το τέταρτο πακέτο παράλληλα. Και θα πρέπει να αποστείλουμε ένα μήνυμα στην Επιτροπή ότι δεν μπορεί κανείς ε, να θέσει σε ισχύ τέτοιους ε, κανονισμούς, να προωθήσει δηλαδή την εφαρμογή τους προς το τέλος μιας θητείας, γιατί αν το προωθεί κάτι τέτοιο κανείς θα έχει τις δυσκολίες που είχαμε και με το τέταρτο ε, πακέτο σιδηροδρομικών μεταφορών, με το πακέτο για τον ενιαίο ευρωπαϊκό ουρανό και γενικότερα ό,τι συνέβη και στο τέταρτο πακέτο το ίδιο ισχύει και για το πακέτο των ε, ε, λιμένων. Στο Στρασβούργο θυμόσαστε οι λιμενεργάτες ότι διαδήλωσαν και αυτή είναι η δεύτερη φορά που μου έπεσαν δακρυγόνα, που μου έριξαν δακρυγόνα. Και το δεύτερο πακέτο για τους λιμένες στη συνέχεια είχε απορριφθεί. Άρα η Επιτροπή δεν, δεν προέβαλε ένα τρίτο παρόμοιο πακέτο, αλλά ένα πακέτο το οποίο δεν ε, σχετίζεται με τις ε, εμπορευματομεταφορές. Ίσως είμαι κάπως ε, αργός, αλλά αν βγάλει κανείς το κάργο δεν καταλαβαίνω πώς μπορεί να προωθήσει ένα πακέτο των λιμένων σε σχέση με τη διακίνηση δηλαδή των φορτίων. Αυτό που έχει σημασία είναι αν βγει βυθοκόρηση, αν βγει αυτή η διακίνηση, τότε δεν παραμένει τίποτα από το αρχικό σε σχέση με τη διαφάνεια, χρηματοοικονομική διαφάνεια ή τη γενικότερη, τις γενικότερες κατευθυντήριες γραμμές αυτών που προωθεί η Επιτροπή. Ε, γι' αυτό νομίζω ότι αν αναστείλουμε τη διαδικασία, δίνουμε την ευκαιρία στην Επιτροπή να αποσύρει αυτό το τμήμα του πακέτου και κατανοώ ότι ίσως θα, δεν θα ήθελα να γίνει μία ε, δεύτερη ε, επαναστατική κίνηση από τους ε, λιμενεργάτες ή έντονη αντίδραση. Από ό,τι κατάλαβα δεν υπάρχει συμφωνία ούτε μεταξύ των βουλευτών. Ο κύριος Φλέκενστάιν έφυξε το βασικό σημείο, δηλαδή τις υποχρεώσεις ε, των δημόσιων επιδοτήσεων. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να κάνει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού σε αυτό το τομέα των κρατικών επιδοτήσεων. Και αν στην επόμενη θητεία με ενδιαφέρει κάτι, είναι να παρακολουθήσουμε τη δράση της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού και πώς αντιμετωπίζει τις κρατικές επιδοτήσεις, γιατί είναι ένας ε, κομβικός ε, τομέας που τους απασχολεί και θα πρέπει και εμείς να το γνωρίζουμε και να το παρακολουθούμε. Νομίζω λοιπόν ότι η απόφαση ήταν απόλυτα σωστή Γι' αυτό αποφασίσαμε να μην δώσουμε συνέχεια σε αυτό το θέμα. Θα δούμε τι θα αποφασίσει το επόμενο κοινοβούλιο. Ε, ο κύριος Λογοθέτης όμως, για λόγους εφταξίας και δημοκρατίας, θα μας πει ποια είναι η άποψη της Επιτροπής και μετά θα επανέλθει ο κύριος Φλέκενστάιν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε και κύριοι. Αντιλαμβανόμαστε ότι ίσως να είναι η τελευταία συζήτηση επί αυτής της πρότασης αυτή την θητεία. Γι' αυτό θα ήθελα να θίξω ορισμένα σημεία. Θα ήθελα να ευχαριστήσω καταρχάς εκείνους που εκτίμησαν το έργο της Κομισιόν και που απευθύναν πολύ ευγενή λόγια προς το μέρος μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να πω ότι καταλαβαίνουμε τα θέματα που αντιμετωπίζει η Επιτροπή Μεταφορών. Το θέμα είναι πολύ βαρυφορτωμένο. Και αυτό εξηγεί γιατί δεν ήρθαμε πιο νωρίς με την πρότασή μας. Το 2007 είχαμε ε, τις μη περιοριστικούς νόμους με το ανακοινωθέν της Κομισιόν. Το 2009 η Κομισιόν άλλαξε και αρχίσαμε να αναλύουμε τι ε, πρόκειτο να συμβεί. Και αυτό πήρε χρόνο. Κάναμε εντελεχείς, μελέτε, μελέτες, κάναμε πολλές αναλύσεις, επισκέψεις, μιλήσαμε με τους υπεύθυνου του κλάδου, είχαμε μεγάλες διαβουλεύσεις. Γι' αυτό πήρε χρόνο να εξισορροπήσουμε το τι έπρεπε να γίνει ανάμεσα σε μη νομοθετικά και νομοθετικά μέσα. Και το 2011 ανακοινώσαμε την αναθεώρηση της πολιτικής λιμένων. Άρα σας παρακαλώ να ε, το δείτε ως το επόμενο βήμα σε έναν αναπόφευκτο τρόπο λειτουργίας. Ήταν μια τόσο σημαντική πρόταση που δεν θα έπρεπε να γίνει με κανένα τρόπο βεβιασμένα. Θα πρέπει να έχετε αντιληφθεί και αυτό έχει τονιστεί από διάφορα μέλη, ότι αυτή η πρόταση έχει πολύ λίγα κοινά με τις προηγούμενες δέσμες 1 και 2. Έχουμε επικεντρωθεί μόνο σε δύο θέματα όπου πιστεύουμε ότι ήταν επιτακτικό να χρησιμοποιηθεί ένα νομοθετικό μέσο. Όλα τα άλλα που περιγράφονται στην ανακοίνωση για την πολιτική των λιμένων έχουν απομείνει ως μη περιοριστικά μέτρα, άλλα μέτρα στήριξης. Αλλά πρέπει να αντιληφθείτε ότι αυτή δεν είναι μια τυχαία πρωτοβουλία. Είναι ένα κομμάτι του puzzle το οποίο αρχίσαμε να φτιάχνουμε προτείνοντας πρώτα απ' όλα ε, τα μέτρα ε, υποδομής που είχατε όλη την ευτυχία και αισθανόμαστε όλοι περήφανοι ως Ευρωπαίοι όταν βλέπουμε ότι ε, είχαμε τις κατευθυντήριες δραγμές για τα ΔΕΔ και τη χρηματοδότηση που έχουν δοθεί για τα διευρωπαϊκά δίκτυα μεταφορών. Γι' αυτό έχουμε και την οδηγία για τις παραχωρήσεις, για τον κοινωνικό διάλογο Όλα τα κομματάκια του πάζολ τώρα μπαίνουν στη θέση τους και αυτά τα δύο μικρά σημεία, πρόσβαση στην αγορά και οικονομική διαφάνεια, είναι τα δύο, δύο κομματάκια που έλειπαν για να κλείσουμε ε, αυτή την εικόνα γιατί ε, προσφέρουμε αυτό σε ένα μεγάλο τομέα ανάπτυξη στην Ευρώπη, δηλαδή τα λιμάνια. Και γι' αυτό αποφασίσαμε να το προτείνουμε παρόλο που είμαστε και στα τελικά στάδια της θητείας αυτής, ε, ενισχύοντας τα ε, δυνατά σημεία των διευρωπαϊκών δικτύων. Θα δώσουμε 26 δις ε, και το κοινό της Ευρώπης θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να ξέρει υπό ποιες συνθήκες θα χρηματοδοτηθούν αυτά τα κομμάτια της υποδομής. Καταλαβαίνουμε ότι ναι, δεν υπήρξε αρκετό χρόνο για αρκετά θέματα. Υπήρχαν διστάμενε απόψει. Το βλέπουμε αυτό και το αντιλαμβανόμαστε πλήρω. Προσπαθήσαμε με την οδηγία των παραχωρήσεων που έκλεισε το κενό εγκαίρως, ε, εγκρίθηκε στα μέσα Ιανουαρίου από εσά εδώ και τώρα ε, ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει σε αυτό τον τομέα. Ε, σε ό,τι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις είχαμε μια ειδική ακρόαση και θα ήθελα να ευχαριστήσω την Επιτροπή που διοργάνωσε αυτή την ακρόαση. Σε αυτή την ακρόαση έγινε σαφές ότι υπάρχουν διάφορες λύσεις. Πρώτον, η νομολογία. Δεύτερον, είναι με τις εξαιρέσει και τρίτον, με ειδικέ κατευθυντήρες γραμμές. Αυτό που θέλω να σας πω αυτή τη στιγμή είναι ότι ό,τι και αν κάνουμε, όποια λύση και αν ακολουθήσουμε στο θέμα των κρατικών ενισχύσεων, η διαφάνεια είναι προαπαιτούμενο. Αν θέλουμε εξαίρεση, ε, θα πρέπει να υπάρχουν βασικά στοιχεία για τις δαπάνες. Αν θέλουμε να ακολουθήσουμε την ομολογία, θα πρέπει να κριθεί ανάλογα με τα γεγονότα. Αν θέλουμε κατευθυντήρες γραμμές, αυτό θα ε, κτιστεί επάνω στα γεγονότα. Και αυτός ο κανονισμός ε, αυτό που κάνει δίνει τα μέσα σε όλες τις αρχές, τις εθνικές, τις ευρωπαϊκές αρχές να εξακριβώσουν τα γεγονότα. Αν θέλει κανείς να ανεξαρτήτως του πού θέλει να πάει κανείς, πρώτα απ' όλα πρέπει να ανοίξει μία πόρτα για να βγει έξω. Αυτό κάνουμε με αυτόν τον κανονισμό. Αυτή η διαφάνεια ανοίγει την πόρτα προς οποιασδήποτε άλλες πρωτοβουλίες. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει με τις κρατικές ενισχύσεις, αυτό είναι το πρώτο και απαραίτητο βήμα που πρέπει να αναλυφθεί. Δηλαδή δεν πρέπει να περιμένουμε μέχρι να ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα μιας μακράς διαδικασίας, αλλά να κτίσουμε επάνω σε αυτό που έχουμε αυτή τη στιγμή στη διάθεσή μας. Αναφερθήκατε στο ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο στάλει και τώρα ε, λόγω του αριθμού γνωστοποιήσεων που έχει λάβει η Κομισιόν, που είναι πολύ μεγάλος. Αυτός είναι ο λόγος. Επίσης, διότι ο κλάδος ζητάει επίμονα να έχει κατευθυντήριες γραμμές και γι' αυτό θα πρέπει να εξακριβώσουμε τα γεγονότα. Γι' αυτό στάλει και τώρα το ερωτηματολόγιο. Λέτε ότι είναι ατυχές. Εμείς λέμε ότι είναι φυσιολογικό. Θέλουμε ε, να ζητήσουμε από την Κομισιόν να κάνει κάτι, η Κομισιόν θα πρέπει να δει τα γεγονότα. Γιατί πρέπει να το κάνει, με ποια, σε ποια βάση πρέπει να το ε, διεκπαιρεώσει. Το πιο θετικό σημείο αυτής της συζήτησης είναι ε, ότι αυτό, αυτή η θητή, αυτό το σώμα, θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Επιτροπή σας και τον Ισχύτη, έχει δώσει λύσεις σε ορισμένα ζητήματα που εμείς εντοπίσαμε, που εντοπίστηκαν στον κανονισμό. Ε, ορισμένα πράγματα δεν ήταν σαφή, ίσως ε, ε, προτείναμε κάπως μια διατύπωση. Η δουλειά που κάνατε εδώ ε, ε λεύκανε ορισμένα σημεία, διευκρίνησε σημεία και ο εισηγητής τα έχει σημειώσει. Έχετε διευκρινίσει θέματα όπως η διαφάνεια, ε, τα τέλη, την εποπτεία, την μείωση του διοικητικού άχθους. Όλα αυτά έχουν διευκρινιστεί και ξεκαθαρίσει και αν συνεχίζαμε θα είχαμε καταλήξει σίγουρα σε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα. Εγώ αποκομίζω από εδώ ότι σίγουρα θα ε, έχουμε ένα πολύ ενδιαφέρον ε, θέμα προς συζήτηση με την επόμενη θητεία και να είστε βέβαιοι ότι η Κομισιόν θα διατηρήσει αυτό που έχουμε εδώ μπροστά μας και μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε την επόμενη προσέγγιση που θα ακολουθηθεί ε, από το ε, κοινοβούλιο στη συνέχεια. Στο μεταξύ, οι συνάδελφοι από το Συμβούλιο θα συνεχίσουν με την εξέταση της πρότασης και σας διαβεβαιώ ότι ε, λαμβάνουν το έργο που γίνεται σε αυτή την Επιτροπή υπόψη τους και έτσι όταν επανέλθουμε στην επόμενη θητεία ελπίζω να έχουμε ένα καλό κείμενο μπροστά μας και από το Συμβούλιο έτσι ώστε να μπορούμε να δουλέψουμε σε συνεργασία προς μια ε, γρήγορη ε, πύληση αυτής της πρότασης που υποστηρίζεται από την πλειοψηφία αυτών που εκφράστηκαν σήμερα. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Γιατί επικρατεί ομοφωνία σε πολλά σημεία είμαι βέβαιος ότι και στην εμφυτεία θα ξεκινήσουμε όχι από το μηδέν, αλλά από εκεί που σταματούμε σήμερα και που διακόπτουμε σήμερα. Δεύτερο. Θέλω απλώ να σας ενημερώσω για τα πρακτικά αυτά που είπα και νωρίτερα, ότι έχω συζητήσει πολύ διεξοδικά με τον κύριο Κουμουτσάκο, μια και δεν μπορεί κανείς να τοποθετηθεί εκ μέρους του ΕΛΚΕΡ να το πράξω εγώ ε, συμφωνούν και το κάνω ως δημοκράτης. Καλώς λέει ο κύριος Σίμψον. Κανονικά θα έπρεπε να ανακοινώσω πότε θα γίνει ψηφοφορία, αλλά ψηφοφορία γιοκ. Και έτσι προχωρούμε και κλεισμένων των θυρών πλέον. Παρακαλώ να αποχωρήσουν όσοι δεν έχουν εργασία για να ενημερωθούμε για τους τρομερείς διαλόγους.